παρουσίαση της εκθέσεως της κυρίας Στάουνερ σχετικά με το σχέδιο δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα ενιαίο πλαίσιο ελέγχων. Τον λόγο έχει η εισηγήτρια για τέσσερα λεπτά. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η βασική αρχή των αποτελεσματικών εσωτερικών ελέγχων είναι και από τις σημαντικότερες αρχές για τα δημοσιονομικά, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και που οφείλει να τηρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποτελεσματικός και γνήσιος έλεγχος προωθείται και ζητείται και από το Ελεγκτικό Συνέδριο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουν γίνει κατ' επανάληψη προσπάθειες, έχουν γίνει επίσης προτάσεις από πλευράς Ελεγκτικού Συνεδρίου, συστάσεις δηλαδή, ώστε τα χρήματα του προπολογισμού να δαπανώνται με τρόπο μετρημένο και φρόνιμο. Ωστόσο, παρόλα αυτά, όλα αυτά τα χρόνια δεν κατέστη δυνατόν το ελεγκτικό συνέδριο να δώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωση θετική αξιοπιστίας. Θυμίζω μόνο τα συμβάντα σε σχέση με ανομαλίε που σημειώθηκαν στην εκτέλεση του προγράμματο Λεωνάρδο πριν από λίγα χρόνια. Επίση, σε άλλου τομεί προγραμμάτων σημειώνονται προφανεί ανομαλίες και υπάρχουν και υποψίες απατών. Τον Ιανουάριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε εν τέλει σχέδιο δράσεως για την δημιουργία εσωτερικών, ολοκληρωμένων εσωτερικών ελέγχων πάλι με τον στόχο να επιτύχει να λάβει θετική δήλωση αξιοπιστίας από το ε, ελεγκτικό συνέδριο. Εν προκειμένου και όπως άλλωστε διαλαμβάνεται και στην έκθεσή μας έχουν γίνει πράγματι προσπάθειες από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπιστώνει ότι η εκτέλεση των μέτρων καθυστερεί σημαντικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει λοιπόν να επιταχύνει την υλοποίηση των μέτρων αυτών και μάλιστα σημαντικά εφόσον επιθυμεί να έχει θετικό αντίκτυπο σε προσεχώς στις εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου έτσι ώστε και οι ευρωβουλευτές να μπορούν να δώσουν με ίσχυη τη συνείδησή τους την απαλλαγή. Δεν θα επισέλθω στις λεπτομέρειες της μη ικανοποιητική εφαρμογής των μέτρων, αλλά τονίζω ότι είναι ακόμα περισσότερο απαραίτητα τα μέτρα ελέγχου διότι για να δοθούν δήθεν ταχαίως οι βοήθειες εν ώψη της κρίσης έχουν μειωθεί, έχει μειωθεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησεως. Γνωρίζουμε όλοι ότι όλα τα μέτρα, ιδίως στον τομέα των διαρθρωτικών ταμείων, λαμβάνονται και εκτελούνται σε συνδυασμό με τι χώρε μέλη. Κάτι το οποίο είναι λογικό και σκόπιμο για να εξασφαλίζει τη σκοπιμότητα των δαπανών. Από την άλλη μεριά όμω, προκαλεί αρκετά σημαντικά προβλήματα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γνωρίζουμε εδώ και χρόνια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την ενέργεια τέτοιων ελέγχων δεν μπορεί πάντοτε να δρά όπω ίσω θα ήθελε και όπω το επιβάλλουν οι αρχέ που επιβάλλει το ελεγκτικό συνέδριο ιδιαίτερο, ιδιαίτερα στις αιτήσεις συνόψεις για τη διαχείριση των πόρων στο εθνικό επίπεδο και που έγιναν για πρώτη φορά υπολήθηκαν τα σχετικά έγγραφα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρώτη φορά στις 15 Φεβρουαρίου 2008 το Κοινοβούλιο δεν μπόρεσε να αποκτήσει ολοκληρωμένη εικόνα διότι τα έγγραφα δεν δίνουν συγκεκριμένα κριτήρια. Έτσι λοιπόν στην έκθεσή μας που ψηφίστηκε ομοφόνος από την Επιτροπή Προϋπολογισμών, ζητούμε από τις χώρες μέλη να είναι πλήρη τα δεδομένα που υποβάλλουν και να είναι και επαληθεύσιμα. Και ζητούμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει σοβαρά τις αρχές αυτές και την ανάγκη τήρησής τους και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Το λόγο λαμβάνει ο Επίτροπος Μπαρό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Στάουνερ για την έκθεσή της και το Κοινοβούλιο για τον επικοδομητικό διάλογο που διεξήχθη από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε ένα σχέδιο δράσεως για μια θετική δήλωση αξιοπιστίας. Σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φρονεί ότι η δήλωση εξοπιστία που δόθηκε το λεκτικό συνέδριο για το 2007 είναι η καλύτερη δήλωση που επετεύχθη ποτέ. Το σχέδιο δράσεως συνέβαλε σε αυτή την βελτίωση. Λοιπόν, έχω τη χαρά να σε ενημερώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε την υιοθέτηση τη πρόσφατη τελευταία εκθέσεω τη όσον αφορά την επιτευχθήσα ε, πρόοδο στι 3 Φεβρουαρίου θα δοθεί. Όπω ζήτησε στην εκθεσή τη η κυρία Στάουνερ, αυτό θα σε επιτρέψει να λάβετε υπόψη στο ψήφισμα διάφορε πτυχέ. Η ανακοίνωση τη 3 η Φεβρουαρίου, τη δική μα ανακοίνωση, παρουσιάζει μια πρώτη αξιολόγηση των συνεπιών του σχεδίου δράσεω μέχρι τι 31 Δεκεμβρίου 2008 συμπεραίνει ότι σημαντικέ πρόοδοι επετεύχθησαν κατά τη διάρκεια τη θητεία τη παρούση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να παραθέσω κάποια σημεία όσον αφορά την απλούστευση. Ε, σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας, ποιο είναι πιο εύκολο να εφαρμοστούν και πιο ευληπτή, αυξήθηκε η εκτέλεση 25% του προπολογισμού. Στα πλαίσια του σχεδίου οικονομικής ανακάψεως προτείνουμε και άλλα μέτρα πλούστευσης, κυρίως για τα διευθυντικά ταμεία. Το ελεκτικό συνέδριο διαπίστωσε μια βελτίωση όσον αφορά τη σαφήνεια και την αξιοπιστία των ετησίων εκθέσεων δραστηριότητα των υπηρεσιών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που συμπεριλαμβάνονται στη δράση 3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσε τι οικονομικέ διορθώσει πράξης 11 όσον αφορά τα εθνικά ταμεία το 2008. Ένα ποσό ενός δις 500 εκατομμυρίων ανεκτήθη εν συγκρίση με ένα ποσό που ανεκτήθη το 2007 που ήταν 288 εκατομμύρια. Η Υπηρεσία Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει και περισσότερο κοινέ προδιαγραφέ όσον αφορά τι μεθόδου ελέγχου. Επιτυχάνεται καλύτερο συντονισμό και γίνεται καλύτερη διαβίβαση των αποτελεσμάτων. Και το διοικητικό άκθο μειώθηκε και εκμεταλλευόμαστε καλύτερα τα αποτέλεσματα των ελέγχων. Θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο τα κατημέλη για τις κοινέ δράσεις, δράση παριθμών 5 και για δεύτερη φορά λάβαμε την ετήσια σύνοψη των ελέγχων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει τις δράσεις της καθώς και άλλες πρωτοβουλίες με σκοπό την βελτίωση του ελεγκτικού πλαισίου. Η έκθεση της κυρίας Στάουνερ υπογραμμίζει τον βασικό ρόλο που έχει η έννοια του ανεκτού κινδύνου όσον αφορά μελλοντικές βελτιώσεις. Αυτή η έννοια έχει στόχο να καθορίσει σε πολιτικό επίπεδο την αποδεκτή ισορροπία μεταξύ αποτελεσμάτων και κόστους των ελέγχων. Είναι προφανές ότι μηδενικό ποσοστό σφάλματος είναι κάτι ανέφικτον και θεωρείται λογικό ότι ανάλογα με το κάθε πεδίο ποικίλει το ποσοστό σφάλματος. Η συζήτηση διοργανική όσον αφορά αυτή την έννοια συνεχίζεται βάσει της πρόσφατης ανακοινώσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Αντιπρόεδρος Κάλλας είχε τη δυνατότητα να μιλήσει αυτό το θέμα μήνα Ιανουάριο στο Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία της εν λόγω πρωτοβουλίας η οποία θα επιτρέψει στην αρχή της απαλλαγής να εκτιμήσει καλύτερα την ποιότητα της αξιολογήσεως του κινδύνου, ε, τη μέθοδο αυτή που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην τελευταία έκθεση βλέπετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε τις διάφορες δράσεις της. Το ελεκτικό συνέδριο θα κάνει τη δική του εκτίμηση και τις, τον αντίκτυπο που έχουν οι, κάθε, οι διάφορες δράσεις στην ετήσια έκθεση του 2008. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Στάουνερ για την έκθεσή της που είναι μια παρακίνηση προς βελτίωση του ε, λογιστικού μας πλαισίου. Έτσι περαιτέρω μάλλον. Σας ευχαριστώ κυρία μου. Äh, ευχαριστώ. Η ψηφοφορία προβλέπεται αύριο. Ακολουθεί η σύντομη παρουσίαση της εκθέσεως της κυρία Σάλ για την ακαιρεότητα των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας ηλεκτρονική συνδεση Η συγκίτρια, τέσσερα λεπτά. Er Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι υπερήφανη